Good morning. Please, could we, could we start this meeting now as swiftly as possible? Take your seat. Καλημέρα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Καθίστε και ξεκινάμε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, θα ξεκινήσουμε με την αναβολή του 25 και άρα η αυριανή θα αρχίσει στις 9.45 με ακρόαση περί των ε, ενδοκρινικών διαταραχτών. Τα πρακτικά Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έχουν κυκλοφορήσει και ε, εφόσον δεν έχουν υπάρξει αντιρρήσεις εγκρίνονται. Να σας ενημερώσω ότι θα γίνει μια σημαντική αλλαγή στη γραμματεία. Είναι, είναι η Ναταλία Παπαστεριάδο που δουλεύει εδώ από το 2013 θα φύγει από τη γραμματεία μας και θα κινηθεί προς την ΕΝΒΗ. Ε, είμαι βέβαια ότι η εμπειρία της ε, από αυτήν εδώ την Επιτροπή θα αποδειχθεί πολύτιμη και ότι δεν θα διασκεδάσετε τόσο στην ΕΝΒΗ όσο εδώ. Ναταλία, ήσασταν πυλώνα τη γραμματεία μα και ε, ήσουν πάντα πολύ αποτελεσματική. Χάρηκα την ευγένειά σου ε, και τη, χιούμορ σου και τη φιλία σου και γι' αυτό θα είμαι πάντοτε ευγνώμων. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το τεράστια δουλειά που έκανες στη διάρκεια αυτών των ετών και γιατί πάντοτε ερχόσουν ε, σε επαφή μαζί μου και τους υπόλοιπους με ιδιαίτερα καλό τρόπο. Φεύγεις από την Επιτροπή, αλλά η φιλία θα παραμείνει. And there are no other business. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό το θερμό μου όλο χειροκράτημα στην Αταλία και να μας θυμάσαι. Όχι μόνο με σύγχυση, αλλά και με χαρά. Που και που. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τώρα. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Όλοι έχετε τις, ψηφοφο... τις κάρτες σας. Βάλτε τις στη σχισμή και πάμε στη γνωμοδότηση για την έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τροπολογία 1 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ναι, αν πρέπει να επιβιώσετε, φανταστείτε εγώ ε, που είμαι εδώ συνέχεια. Τρέξε, τρέξε στη θέση σου και βάλω και την κάρτα σου στο μηχάνημα, λέει η πρόεδρος. Και ξεκινάμε. This is by hand, so who is in... Μάλιστα, τώρα δυνατά τη χειρός. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της τροπολογίας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ναι, δεύτερο τμήμα είπαμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. in favor. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, πρώτο τμήμα, ναι, ναι, πρώτο τμήμα, υπέρ, games, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Vote is... Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is still open. Ψηφίστε παρακαλώ. And now the vote is closed. Και τώρα τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Ε, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. And Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Χρειάζεται να υποδείξετε ή αν είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ, ποιοι είστε, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός. Same voting pattern. 13. Για την 13 ψηφίζουμε. Άρχεται και τέλος. Απορρίφθηκε. Είδατε όμως είναι ίσα ίσα, πρέπει να το ελέγξω. 15 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, ξέχασα τη 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 16 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Α, αυτό καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική 8, υπέρ. Κατά αποχές, γίνεται. Πάμε στην τροπολογία 25, δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά. Τέλος της πληροφορίας. Ε, Τροπολογία 29. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ, πρώτο τμήματος, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 44 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίθηκε. Τροπολογία 40 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Ε, και κοιτάξτε πάλι, ισοπαλία, ισοψηφία, απορρίπτεται. 45. Ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 45 δεύτερο τμήμα. The uh, vote is... We close the vote. Τέλος. Ωραία, απορρίφθηκε. 46. Δύο τμήματα. το πλήρες κείμενο. Ποιο είναι υπέρ. 46, the first part. The first part. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει και πάμε στη 47 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χρειάζεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά Let's open the vote to check. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο της τροπολογίας 55. Και τώρα τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Έχουμε λοιπόν κάποιους εδώ που εξαρτώνται από μένα. Λοιπόν. 48. Δεύτερο τμήμα θα ψηφίσουμε πρώτα όμως. Το δεύτερο τμήμα του 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέσε δεν εγκρίθηκε, απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές ε, καλύτερα να επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν πέρας και απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Πολύ στενά τα αποτελέσματα σήμερα. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως ε, είναι η ίδια πλειοψηφία. Θα ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά επί της 53. Πέρας. Α, τώρα εγκρίνεται όμως. Ευτυχώς που το τσεκάραμε. 54. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές. εδώ πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 53. Συγγνώμη, 63. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη πάλι με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση βεβαίω να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί με ισοψηφία. Είμαστε στην τροπολογία 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία από τις 66. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα της 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές ε, και εδώ δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Τροπολογία 51 έχει αποσυρθεί, τροπολογία 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε πολύ ωραία τροπολογία 75. Πέρασε και απερίφθη. 76 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, έχει αποσυρθεί. Στο δεύτερο τμήμα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε το αποτέλεσμα αυτό. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. 77 είναι η τροπολογία. Πέρας και απερίφθη. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική τροπολογία τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ή e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ας ψηφίσουμε επί της ονομοδοτήσεως στο σύνολό της και αυτό θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα Στη δεύτερη ψηφοφορία, προφορική ερώτηση, θα ψηφίσουμε λοιπόν επί του κειμένου της προφορικής ερωτήσεως και θα γίνει η ψηφοφορία με ηλεκτρονική διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now closed. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε λοιπόν και Ολοκληρώσαμε τώρα τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθαν μόνο για την ψηφοφορία. Εάν εγκαταλείψετε την αίθουσα, παρακαλώ πολύ να το πράξετε ησύχως. Χαίρομαι που βλέπω εδώ και μερικά πρόσωπα συναδέλφων που δεν έρχονται συχνά και ελπίζω να τους ξαναδούμε συχνά, να περάσουν ξανά από τα μέρη μας.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 working day, which is going to be long. We are going to finish this afternoon at 6. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε την ε, αναφορά 92 σχετικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. It's Peter Zatmari. And I would be happy to see... Όμως ε, Έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πού βρίσκεται. Α, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πράγματι, η αναφορά αυτή αφορά προβλήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται ε, με την ε, παράκαμψη ε, φορτηγών αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο σε ένα δευτερεύοντα δρόμο που δεν έχει διόδια. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ε, σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, χρέωση στους αυτοκινητοδρόμους και αφορά ακριβώς ε, και τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Η νομοθεσία αυτή δεν επιβάλλει χρέωση από πλευράς ε, του κράτους ε, μέλους. Ε, επομένως, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει με απολύτως ελεύθερο τρόπο εάν θα χρεώσει ή όχι και πόσο θα χρεώσει την χρήση των δρόμων. Μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ένα ανώτατο όριο στην χρέωση αυτή. Ε, εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση ανάμεσα σε χρήστες οδικού δικτύου. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση ιδιαιτέρωση στην Ισπανία όπου ε, υπάρχουν παρόμοιες ε, υποδομές ε, ε, κάποιοι δευτερογενεί δρόμοι οι οποίοι γίνονται πολύ ελκυστικοί ε, για τους χρήστες. από την άλλη πλευρά βεβαίως και αυτό θα είναι και η κατακλίδα τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητα έτσι ώστε να εξεύρουν τα κατάλληλα κυκλοφορικά μέτρα τα οποία θα μέτρα για ελέγχου της κυκλοφορίας ε, και ε, γνωρίζουμε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή ε, στην Ισπανία υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται με μείωση της χρέωσης στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έτσι έχουν τα πράγματα, ε, δεν έχουμε άλλη αρμοδιότητα. Εδώ μιλάμε για αρμοδιότητα του κράτους μέλους ε, να διευθετήσει την ε, κυκλοφορία στους δρόμους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά μιλήσατε μόνο επί του προκειμένου. Βαλέν, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η χρέωση των, αυτοκινητοδρόμου ε, αυτοκινητοδρόμους ε, είναι σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση και συντήρηση των υποδομών. Υπάρχουν λοιπόν κάποια, κάποια αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πολύ από ιδιαίτερα ε, βαρέα οχήματα. Από την άλλη πλευρά πολλά βαρέα οχήματα πηγαίνουν σε δευτερογενείς δρόμους για να αποφύγουν την πληρωμή των δίων. Ε, αυτό ε, βεβαίως σημαίνει ότι το εξωτερικό κόστος ε, μπορεί να αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου καλούνται τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την οδική χρέωση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας αυτής ε, αφορά μονάχα συγκεκριμένους αυτοκινητοδρόμους. Απ' την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν πώς ε, θα δημιουργήσουν τι απαραίτητε δομέ και πώς θα διαχειριστούν την κυκλοφορία και πώς θα δημιουργήσουν παρακαμπτήριες από τους κεντρικούς αυτοκινητοδρόμου σε άλλου. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. Η διαχείριση ε, των, ε, των οδών και των ε, παρακαμπτηρίων αφορά μονάχα τα κράτη-μέλη και είναι δική τους αρμοδιότητα. Ε, λαμβάνοντα ε, υπόψη όμως ε, την χάρτα για την οδική ασφάλεια, μπορεί η Κομισιόν να μας πει κάποια στοιχεία τα οποία να σχετίζονται με το τι θα συμβεί μετά από το 2020 και όταν θα αρχίσει να ισχύει το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια και αν εκεί προβλέπεται λύση για κάποια προβλήματα σαν αυτά που συζητούμε σήμερα. Θα πρέπει κατά την άποψή μου λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να λάβουμε ε, πιο συγκεκριμένες πληροφορίες από πλευράς της Κομισιόν για τα θέματα τα οποία έθεσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Νάκ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Εθνικός Αυτοκινόδρομος 1 ε, μου είναι πολύ γνωστός γιατί τον έχω περπατήσει τον έχω οδηγήσει πολλές φορές. Είναι ένας όμως αυτοκινητόδρομος ε, με πολύ μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων και έχει δίπλα του ε, τον API ε, AP1 που είναι η συνέχεια του άξονα η EO5 του ευρωπαϊκού άξονα. Ε, ε, στη μία περίπτωση υπάρχουν διόδια ε, ήδη από το 1994. Μια παραχώρηση στην οποία ο παραχωρησιούχος είχε επιμήκυνση του συμβολέου. Εδώ μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο που έχει τεράστιο ποσοστό ατυχημάτων, αλλά και γενικά το ξέρουν όλοι στην Ισπανία και υπάρχουν, είναι, είναι η σύνδεση με τη Γαλλία και τα ατυχήματα είναι πάρα πολλά. Είναι σαφές ότι η αρμοδιότητα τα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ. Έχουμε επίσης τον 13-15 του 2013, Δεκεμβρίου μάλιστα του 2013, ε, όσον αφορά τους προσανατολισμούς για την ανάπτυξη οδικών ε, μεταφορών. Και εδώ μιλάμε ε, για την AP1 που αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο και επομένως αυτό το κείμενο λέει για να εγγυηθεί η διεθνής κινητικότητα των εμπορευμάτων και των επιβατών θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος και να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να μην υπάρξουν πλέον μποτιλιαρίσματα, να μην υπάρχουν σημεία δηλαδή συμφόρησης. Εδώ τα προβλήματα προκύπτουν ακριβώς λόγω της συμφόρησης. Εδώ επίσης έχουμε και κάποια μελέτη η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την λήψη μέτρων που υποτίθεται υποτίθεται ότι θα μείωναν κατά 50% μάλιστα τα ατυχήματα, τίποτα τέτοιο βέβαια δεν συνέβη. Ε, υπό την Μαλτέζικη Προεδρία έγινε μια προσπάθεια ε, να προχωρήσει το θέμα της οδικής ασφάλειας. Εδώ μιλάμε επομένω για θέμα το οποίο σχετίζεται σαφώς με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επομένως δεν πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά γιατί εδώ μιλάμε για πολίτες οι οποίοι υποφέρουν από τα σημεία συμφόρησης ε, αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Και επίσης μιλάμε για την AP1 η οποία εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Solidad, welcome back. Καλώς ήρθες Σολεδάδ, λέει η Πρόεδρος ε, ξανά. Χαίρομαι που είσαι εδώ και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Bueno, efectivamente. se trata de Πράγματι, εδώ μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο με διόδεα ε, που ανακαινίζεται ε, υπήρχε μια ε, ε, παραχώρηση για, την, για τα συγκεκριμένα διόδια που δίδηκε σε 20 χρόνια και τώρα πρέπει να ανανεωθεί και εντάσσεται και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση ή με την πολιτεία. Ήδη από το 1995 αναγνωρίζεται ότι ο υψηλός βαθμός, ο ποσοστό ατυχημάτων αυτού του αυτοκινητοδρόμου και του δευτερογενούς αφορά ακριβώς, ε, οφείλεται μάλλον, ε, στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό βαρέων οχημάτων. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, ε, είναι ε, γεγονός ότι είναι καταχρηστική γενικά η πολιτική των αυτοκινητοδρόμων ε, στην Ισπανία. Έχουμε πρόσφατους αυτοκινητοδρόμους που έχουν τεράστια διόδια. Απ' την άλλη μεριά έχουμε άλλους αυτοκινητοδρόμους όπως αυτό που οδηγεί στο Κάντι, θα πούμε που δεν ανακαινίζονται και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στους κατοίκους. Εδώ μιλάμε για, στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, για πολλά χωριά, μικρά χωριά και κομοπόλεις που φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Ε, ωστόσο μιλάμε για χωριά και κομοπόλεις ε, η επικοινωνία μεταξύ των οποίων γίνεται οδικά και είναι απολύτως σημαντική. Αυτό που πρέπει να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο είναι βεβαίως τον Νοέμβριο ε, να ε, μην ανανεώσει το συμβόλαιο και να απελευθερώσει ε, τον, το συμβόλαιο με τον παραχωρησιούχο. Η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη είναι τον 13-15 κάθετος 2013 που αφορά την, την διεθνή μετακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών και που αναφέρει συγκεκριμένα ότι θα πρέπει θα πρέπει να αποφεύγονται ε, τα σημεία συμφόρησης, γιατί ακριβώς από εκεί προκύπτουν τα προβλήματα. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το θέμα, κυρίως γιατί πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο που αφορά και την επιβίωση των ντόπιων αλλά και την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ιτουργκάης. Mm. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω πολύ καλά τον δρόμο αυτό, γιατί είναι πολύ κοντά εκεί που μένω. Μάλιστα λέγεται ο δρόμος των Πορτογάλων, γιατί πολλές φορές ε, διασχίζουν ε, την Ισπανία οι ε, Πορτογάλοι που πηγαίνουν προς την Πορτογαλία ή αντίθετα που έρχονται προς την ε, Γαλλία την ε, ναι, και την Βόρεια Ευρώπη. Αυτός ο δρόμος λοιπόν είναι ένα από τα, μεγάλα μαύρα σημεία που συναντά κανείς στην Ισπανία στο δίκτυο το δικό μας. Ε, περνάνε πάρα πολλά φορτηγά και να θυμίσω ότι περνάνε από εκεί τα φορτηγά γιατί τα διόδια για το συγκεκριμένο εθνική του Μπούργος είναι πολύ πιο ακριβή. Είναι, είναι αρκετά ακριβή σε, σχέ, σε σχέση με άλλους αυτοκινητοδρόμους που έχουμε στην Ευρώπη. η συνάδελφο Καπεθών είχε δίκιο όταν έλεγε ότι θα πρέπει αυτό να μεταβιβαστεί, να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα ε, δύσκολα σημεία που υπάρχουν στην Ευρώπη, στο δικό δίκτυο, στις εθνικές οδούς κτλ. Και, τις εθνικές ε, αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Και μέσα από αυτή την αναφορά θα μπορούσαμε να πάμε και σε άλλες αναφορές μια έκθεση ή, εν πάση περιπτώσει, μια μια, ένα έγγραφο της Επιτροπής Μεταφορών όπου θα εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα. Η Κομισιόν λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει και λέει πως δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας αλλά εθνικής αρμοδιότητας και εδώ θέλω κυρία Πρόεδρε τα δύσκολα αυτά σημεία, τα προβληματικά σημεία των ευρωπαϊκών δρόμων, των ευρωπαϊκών εθνικών οδών, θα έπρεπε να είναι θέμα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τη Επιτροπή Μεταφορών, που συζητούν αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν εγώ είμαι υπέρ του να διαβιβαστεί, πρώτα απ' όλα να μην ανοιχτεί και δεύτερον να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών, αν συμφωνείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Τώρα η επιτροπή μας έγινε ισπανική. Πολύ ωραίο, αλλά και σύνηθες. Ευτυχώς θα ακούσουμε και την κυρία Κρόης. Αλλά <laughs> τώρα σας ζητώ συνάδελφοι, γιατί βλέπω πως όλοι θέλουμε το ίδιο στην ουσία. Να είστε λίγο σύντομοι, γιατί ο χρόνος ε, ε, παίρνει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ζητώ από την κυρία Μιράντα τώρα να πάρει το λόγο όσο γίνεται πιο σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη μου παρέμβαση σε αυτή την Επιτροπή Μεταφορών και θέλω να τονίσω πως το πρόβλημα αυτό όντως θα πρέπει να μείνει ανοιχτό γιατί είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και επηρεάζει τις οδικές μεταφορές. Το, το ποσοστό των ατυχημάτων είναι πολύ μεγάλο. Ε, ε, άρα έχουμε να κάνουμε εδώ με την ασφάλεια του δικού του σιδηροδρομικού και του αεροπορικού δικτύου. Θα πρέπει ωστόσο να κάνουμε και ένα βήμα ακόμα σε σχέση με την ε, διόρθωση των δρόμων και άλλων εθνικών οδών που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι και άλλες εθνικές οδοί που έχουν προβλήματα. Παρακαλώ λοιπόν να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Κυρία Κρόης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπής ΤΡΑΝ και είμαι και συντονίστρια για όλες τις ε, αναφορές που αφορούν το πεδίο των μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά ώστε να δούμε με κάθε λεπτομέρεια αυτό το ζήτημα. Είναι λοιπόν σωστό να μείνει ανοιχτή και για, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτήν εδώ την αναφορά. Θα στείλουμε έκθεση, μάλλον επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας. Και μετά θα στείλουμε και στην Επιτροπή Μεταφορών να ζητήσουμε τη γνωμοδότησή τους. Αυτά μπορούμε να κάνουμε για την ώρα. Ήδη είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Νομίζω καταρχάς ότι θα το διαβιβάσουμε σε άλλη επιτροπή και ε, φυσικά θα πούμε και στους Ισπανούς ότι μας ανησυχεί το θέμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εξαιρετικά. Και πάμε στην επόμενη αναφορά που είναι το σημείο 9 και νομίζω ότι ο αναφέρον δεν, ή αναφέρουσα μάλλον, δεν είναι ακόμα εδώ. Ε, και άρα πάμε στο σημείο 10, τη 224, να την ε, κλείσουμε αυτή και μετά να επανέλθουμε στην 9. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με το σύνδεσμο βουλγαρικών σχολείων Αλοδαπή, φέρει 1.707 υπογραφέ σχετικά με την πρόταση διενέργεια των τελικών σχολικών εξετάσεων σε όλε τι επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, αναφέρουσα είναι εδώ, είναι η κυρία Κόνα Κίεβα. Ε, συγγνώμη δεν προφέρω καλά το όνομά σα. Είστε πρόσδεκτοι λοιπόν εδώ και σα δίνω μάλλον το λόγο για πέντε λεπτά. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, Асоциацията на българските училища в чужбина ви благодаря. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Είμαστε γνώμονες που μας καλέσατε. Προσωπώ τον σύνδεσμο των βουλγαρικών σχολείων στην Αλοδαπή. Η, έκθεση, η αναφορά μας φαντάζει έγινε ενώ ε, γνωρίζαμε περίπου ποια θα είναι η απάντηση, διαβάσαμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα όμως να σας ε, ε, εντυπωσιάσω λέγοντας σας τι δεν ζητάμε με αυτό την αναφορά. Δεν ζητάμε την αναδιοργάνωση, τη μεταρρύθμιση του συστήματος παιδείας ή των πολιτικών περιγλωσσών, είτε την εναρμόνιση, ούτε τίποτα τέτοιο πράγμα που δεν γίνεται και δεν είναι σύμμορφο Προ την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουμε είναι συντονισμός ε, σύμφωνα με το άρθρο 165 τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται αυτό το μέτρο, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει εκατοντάδε χιλιάδε ευρωπαϊκέ οικογένειε, ε, καθώ και τα παιδιά του. Ε, παιδιά τα οποία μιλούν εννέα τουλάχιστον από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση και δεν μιλάμε για την παιδεία εδώ στην πράξη, μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και για την κινητικότητα. Μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία του πιο σημαντικού κεφαλαίου που έχουμε, της νεότητάς μας. Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι και κομμάτι πολύ σημαντικό ε, των δεξιοτήτων των παιδιών μας ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα παιδιά να μαθαίνουν γλώσσες, ωστόσο λόγω μετακίνηση σε μια άλλη χώρα, τα παιδιά μπορεί να μην μπορούν να μάθουν μια γλώσσα ή να συνεχίσουν να μιλούν μια γλώσσα που ήδη μιλούν. Για ένα παράδειγμα, όσοι έρχονται από τη Βουλγαρία, στο σχολείο μαθαίνουν γαλλικά και αγγλικά. Ενώ αν κινηθούν στη Γαλλία ε, μαθαίνουν μόνο μία ξένη γλώσσα, τα αγγλικά, γιατί τα βουλγαρικά δεν μετράνε στο νέο του σχολείο. Δεν διδάσκονται δεν εξετάζονται και στην πράξη το τοπικό σύστημα στέλνει το μήνυμα πως αυτή η γλώσσα είναι περίτη, άχρηστη. Μπορεί κανεί να πει κάτι τέτοιο όμω, ότι μια γλώσσα είναι άχρηστη, ότι τα κράτη-μέλη τη δεν χρειάζονται τη γλώσσα του ότι δηλαδή οι νέοι δεν χρειάζεται να μιλούν τη γλώσσα των άλλων κρατών μελών. Εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε ολοκλήρωση της αγοράς και της, ε, του πολιτισμού μας, αυτή η έλλειψη αναγνώρισης, ε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δυσκολία για, ε, για τις οικογένειες που θέλουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό, εφόσον τα παιδιά τους είναι στο γυμνάσιο. απλά και μόνο επειδή τα παιδιά τους έτσι αγαστερηθούν τη δυνατότητα να ε, μάθουν μια επιπλέον γλώσσα. Και άρα θα υστερούν και στις ε, πανεπιστημιακές τους σπουδές αργότερα. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ε, κάποια αντίμετρα και κάποιες οδηγίες κάποιοι ε, ε, διευθυντέ σχολείων διοργανώνουν ε, εξετάσει. Αυτό συμβαίνει, α πούμε, στη Γερμανία, όπου δέχονται του ελέγχους Η Ιρλανδία επίσης έχει θεσπίσει εξετάσεις σε γλώσσες που δεν διδάσκονται στη χώρα στο τέλος του γυμνασίου και η Ουγγαρία χρησιμοποιεί έναν άλλο μηχανισμό που δέχεται τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά από ευρωπαϊκά κέντρα ελέγχου ε, των, ε, της γνώσης των γλωσσών και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της, ε, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το μέτρο λοιπόν που ζητούμε μπορεί να βασιστεί σε αυτό το κοινό πλαίσιο αναφοράς και το άρθρο 165 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται σε αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει κάποιο είδους μηχανισμός για την αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών ανεξάρτητα από το πώς έμαθαν τις γλώσσες. Δεν ζητάμε καμία εναρμόνιση. Τα κρατημέλη θα αποφασίζουν αν θα κάνουν ευρωπαϊκού επίπεδου εξετάσεις, αν θα διδάσκουν και πώς μέσω συστήματος αναγνώρισης πιστοποιητικών, αν θα έχουν εξοδοτημένα σχολεία κτλ. Εν πάση περιπτώσει για μας είναι διοικητικό το μέσο, μέτρο αυτό, δεν είναι εκπαιδευτικό μέτρο και Όπως είπα, πρόκειται για κάτι που δημιουργεί δυσκολίες για πολλούς από τους μαθητές. Εδώ, μάλιστα σήμερα, έχουμε ε, μια-δυο οικογένειες ε, γαλλοβουλγαρικές που θέλουν να μπορούν να κινούνται εύκολα, ε, θέλουμε να είναι ανοιχτέ οι πόρτες για όλους, ε, θέλουμε και να προστατεύσουμε τα αγαθά, ε, την οικονομία, τη φύση, γιατί να μην προστατεύουμε και τις γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η, η Επιτροπή μας γίνεται βουλγαρική. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Κριστίνα Κάνιχα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Madam Chairman. Good Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίε και κύριοι. Ευτυχής που βρίσκομαι παρέα σας ε, σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Κονακίεβα, την αναφέρουσα, καθώς και όλους όσοι υπέγραψαν αυτό, αυτή την αναφορά, διότι είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Και Αναφερθήκατε στις παρατηρήσεις της Επιτροπής ε, που υποβλήθηκαν στην δική σας Επιτροπή φέτος τον Ιανουάριο και θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω για το τι έχει συμβεί έκτοτε. Αμέσως μετά από τις παρατηρήσεις, της, την υποβολή μάλλον των παρατηρήσεων της Επιτροπής, η πρόταση για αναθεώρηση του πλαισίου κλειδιού για τις δεξιότητες εγκρίθηκε και από την Κομισιόν. Και όπως ήδη έχουμε τονίσει, ένα από τα κεντρικά σημεία αυτής της αναθεώρησης αυτού του πλαισίου δεξιοτήτων, που είναι νομίζω αρκετά γνωστό και αναπτύχθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι η ιδέα του αλφαβητισμού και της μάθησης γλωσσών έπρεπε να αναθεωρηθούν δεδομένες της ε, αποδοχής ότι η γλώσσα της εκπαίδευσης δεν είναι αναπαραίτητος η μητρική γλώσσα κάθε μαθητή. Αυτό είναι κάτι που τώρα το έχει σκεφτεί η Κομισιόν ε, και μάλιστα μας απασχολεί εντόνως. Έπειτα, Επίσης ανακοινώσαμε ήδη τον Ιανουάριο ότι μετά από την ε, συμβολή της Κομισιόν στην διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμποργκ τον περασμένο Νοέμβριο θα γνωρίζετε ίσως ότι η συμβολή της Επιτροπής σε αυτή τη συνεδρία ήταν μια ανακοίνωση που έφερε τον τίτλο «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας μέσω της παιδείας και του πολιτισμού». Αυτή η ανακοίνωση εκθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα επιτευχθεί μια ένας ευρωπαϊκός χώρος παιδείας και πρότεινε μετα, μεταξύ άλλων μια πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συν σύσταση να υποστηριχτεί η, η, γνώση, μάλλον, η μάθηση γλωσσών. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή η αναφορά είναι εξαιρετικά επίκαιρη γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση ε, σύνταξης αυτής της σύστασης για την ε, βελτιωμένη εκμάθηση γλωσσών. Όσον αφορά τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την αναφορά, που είναι περισσότερο διοικητικού τύπου, φυσικά είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι συγκεκριμένο τώρα, αλλά και ξέρω και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τα όρια, τους περιορισμούς των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, Χωρίς να θέλω να αποκαλύπτω τίποτα για το τι θα περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύσταση, μπορώ να σας πω ότι γίνεται λόγος για μια συνολική ε, άποψη για την εκμάθηση γλωσσών. Αυτό πρέπει να δούμε αν τέτοια μέτρα σε αυτά που προτείνονται σε αυτήν την αναφορά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια τέτοια συνολική αναθεώρηση. Υπάρχουν και παράλληλα διάφορες πρωτοβουλίες από διάφορες ομάδες συμφερόντων. Η Κομισιόν προσεκλήθη πριν από κάποιες εβδομάδες στην Επιτροπή των Περιφερειών και σε μια διάσκεψη που διοργάνωσαν οι Ευρωπαίοι σε ολόκληρο τον κόσμο και Μάλιστα νομίζω πως η αναφέρουσα επίσης ε, εκπροσωπήθηκε σε αυτή τη διάσκεψη και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, εκεί διαπιστώσαμε πόσοι πολύ ισχυροί οργανισμοί υπάρχουν στην ε, Ενώση, στην Ευρώπη που στηρίζουν την διδαχή και εκμάθηση των διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των Ευρωπαίων όχι, που όχι μόνο κινούνται εντός Ευρώπη, αλλά γιατί εδώ ε, φυσικά έχει να κάνει αυτό με την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και παγκόσμια, σε ολόκληρο τον κόσμο κινούνται. Οπότε πραγματικά πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη ε, και είμαστε ανοιχτοί, ακούμε όλες τις διάφορες πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένες της δικής σας για να δούμε πόσο μακριά θα φτάσουμε στην πρότασή μας που θα κατατεθεί τον Μάιο αυτού του, αυτής της χρονιάς θα, θα θα δείξει στο τέλος, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε επαφή. Είμαι βεβαίω ότι θα είμαστε σε επαφή σχετικά με όλα αυτά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όντως και βλέπω ότι πολλοί Βούλγαροι συνάδελφοι, αλλά και ένας που δεν είναι Βούλγαρος, ε, θέλει να πάρει το λόγο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι, αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να δώσουμε 1,5 λεπτό στον καθένα. 90 δευτερόλεπτα, το ξέρουμε αυτό από το Στρασβούργο. Ο κύριος Μάλινο θα έχει το λόγο πρώτο. Yes. My time is running up, so... Ναι, τώρα θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος μου. Θα μου δώσετε τα 20 λεπτά που έχασα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την ε, αναφέρουσα κυρίως ε, ε, σε σχέση με την ποιότητα και την ε, σαφή κατανόηση των περιορισμών που αναφέρονται στην αναφορά αυτή. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε πιο φιλόδοξα αιτήματα. Συμβαίνει συχνά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στον αναφέροντα εστιάζοντας στην ίδια ε, κατεύθυνση, λες και δεν έχουν υπάρξει προηγουμένως ε, επαφές αυτό το θέμα λοιπόν είναι κάτι που αφορά την βουλγαρική γλώσσα που είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και ε, αφορά βέβαια επίσης και όλες τις μικρές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι στο αίτημά μας. Δηλαδή, αφενός να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, αλλά επίσης θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τίνουν ιδιαίτερο ευήκονους στα όσα θα ακουστούν εδώ και στα όσα θα διαμειφθούν εδώ και να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό. Έτσι ώστε ε, θα ήθελα επίσης να χρησιμοποιήσω μάλλον και τους εσωτερικούς μας κανονισμού λειτουργίας έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Προτείνω λοιπόν στους συντονιστές της Επιτροπής Αναφορών να συζητήσουν την δυνατότητα υποβολής προφορικού ερωτήματος στην Κομισιόν που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια σχετικά με την δυνατότητα βελτίωσης της εκμάθησης γλωσσών και της αναγνώρισης των, γλωσσικών, των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Αυτό ε, βέβαια είναι θέμα που αφορά την κυρία Ποσκόφη, η οποία είναι εισηγήτρια ε, ε, στην Επιτροπή πολιτισμού και την, ε, και την ε, άλλη συνάδελφο η οποία ασχολείται με την πολυγλωσία γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία χρήσουν συζητήσεως στην Ολομέλεια ε, και βεβαίως και στην Ολομέλεια όπως και τώρα περισσότερο από ποτέ θα βασιστούμε στους διερμηνείς. Ναι, θα μεταφέρουμε το μήνυμα που έχουμε. Μόλις έλαβα μήνυμα ότι έχουμε κάποιον από τις βουλγαρικές αρχές. Μπορείτε να παρέμβετε μετά όμως από τη λήψη του λόγου από τα μέλη μας. Εσείς κύριε Νέκοφ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Να συγχαρώ την κυρία Κονακτσίεβα καθώς και τον Διευθυντή του Βουλγαρικού Σχολείου Βρυξελών. Υποστηρίζουμε την ιδέα να συζητηθεί το θέμα αυτό και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι και σκιώδης εισηγητής για σχέδιο ψηφίσματος για την χρήση περισσότερων γλωσσών στην ψηφιακή εποχή. Και όπως είπα είμαι σκιώδης εισηγητής και θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το θέμα αυτό να ευθυγραμμιστεί, να μπει δηλαδή σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος του Κοινοβουλίου, ώστε το καθεστώς των μικρών γλωσσών να προωθηθεί, γιατί η πολιτιστική ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών, είτε έχουν γεννηθεί στη Βουλγαρία, είτε έχουν γεννηθεί αλλού, ας πούμε στη Βρετανία, είναι σωστό να διαθέτουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους. Και όπως λέει και η κυρία Κονακτσίεβα, η πολυγλωσία είναι σημαντικό στοιχείο του ενεργητικού της ε, Ένωσης. Βεβαίως ε, υπερισχύει η χρήση της Αγγλικής. Αλλά δεν μπορούμε να μετακινηθούμε από τη θέση μας. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν καλά με τα αγγλικά. Στη Βουλγαρία λιγότεροι από 20% των πολιτών κατανοούν τα αγγλικά. Γι' αυτό οι πολυγλωσσικές πρακτικές είναι σημαντικές. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Βλέπω ότι ο κατάλογος γίνεται όλο και μακρύτερος και έχω ήδη 10 εγγεγραμμένους και καθυστερούμε. Κύριε Ράντεφ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όπως είπαν και οι συναδελφοί μου, θεωρώ ότι η αναφορά των βουλγαρικών σχολείων Αλλοδαπής ε, είναι σωστή. Οι περισσότερες χώρες μέλη δεν προβλέπουν τη δυνατότητα να γίνονται εξετάσεις σε άλλες γλώσσες στην, κατά την αποφύτιση από την δευτερεύουσα από τη, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από ορισμένα ε, σχολεία που ε, ε, διδάσκουν γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και αυτό αποτελεί διάκριση σε βάρος των σπουδαστών λόγω ηθαγένειας. Να το αλλάξουμε αυτό, ώστε οι επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες να γίνουν ευρύτερα γνωστές. Και ε, αυτό θα διευκολύνει και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Σας ευχαριστώ. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε στα αγγλικά. Υποστηρίζω τις δύο προτάσεις του κυρίου Μαλινόφ και επομένως σύνταξη επιστολής προς ε, τους ε, αρμόδιους υπουργούς. να σημειωθεί πρώτα τα όσα, να σημειωθούν μάλλον πρώτα τα όσα είπαν τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα συνολική προσέγγιση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για τα συμπεράσματα του Γκέτεμποργκ και για τον κοινωνικό πυλώνα. Στα βουλγαρικά η αρχή νούμερο 1 έχει ως εξής, θα σας τη μεταφράσουμε. Η αρχή αυτή του κοινωνικού πυλώνα είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση και διαβίου εκπαίδευση. Ο κάθε ένας και η κάθε μία έχουν δικαίωμα σε πρόσβαση σε εκπαίδευση καλής ποιότητας και σε διαβίου κατάρτιση που να προσφέρει τη δυνατότητα στο πρόσωπο να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που θα το καταστήσουν ικανό να συμμετάσχει στην κοινωνική ζωή. Και βεβαίω και στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Κύριε Σαντενόφ, παρακαλώ, όλες και όλοι. Γνωρίζουμε ότι συμφωνείτε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τα όσα έχουν πει ήδη οι συναδελφοί σας. Άρα, σα παρακαλώ να είστε πραγματικά συντομότατοι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υποστηρίζετε. Ελπίζουμε μόνο να μπορέσουμε να προσθέσουμε επιχειρήματα, λέει ο κ. Σπυρίνσκι. Αντενόφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, πράγματι, ε, επαναλαμβανόμαστε. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσφέρουμε υποστήριξη στην αναφορά της κυρίας Κοναξίωρα. Διότι, δυστυχώς, αυτές οι λεγόμενες μικρές ευρωπαϊκές γλώσσες υφίστανται διακρίσεις. διότι δεν μπαίνουν μέσα στα διεθνή σχολικά συστήματα και όλο και περισσότερες οικογένειες με παιδιά ε, ε, μετακινούνται και εγκαθίστανται σε άλλες χώρες μέλη όπως έχουν το δικαίωμα από τις συνθήκες θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχαν και τη δυνατότητα να μαθαίνουν τη γλώσσα τους. Είναι σαφές ότι το κοινό πλαίσιο αναφοράς και τα εφιστάμενα κέντρα εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα, να κινηθούν όλα προς την ίδια κατεύθυνση, διότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι μια ανοιχτή, ανεκτική Ευρώπη. Εμείς να στείλουμε την αναφορά και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, διότι θα πρέπει να φροντίσουν να άρουν τις διακρίσεις αυτές σε βάρος των παιδιών. Κορομποσέφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω κάποια επιχειρήματα ακόμη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ανεξαρτήτως του πόσες γλώσσες μιλεί κάποιο πρόσωπο, η γνώση της μητρικής γλώσσας έχει κρίσιμη σημασία. Στο βουλγαρικό σχολείο των Βρυξελών υπάρχουν 50 παιδιά στην πρώτη τάξη του δημοτικού και μέχρι να φτάσουν στο τέλος όμως της σχολικής εκπαίδευσης μένουν 5 διότι δεν έχουν κανένα κίνητρο να συνεχίσουν να διδάσκονται στην ε, μήτρικη τους γλώσσα. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθαρά βουλγαρικό θέμα, είναι ευρωπαϊκό θέμα. Προσπαθήσαμε να το επιλύσουμε διμερώς, μιλώντας και με διάφορες άλλες χώρες μέλη. Αλλά η προσπάθεια αυτή είναι εξαντλητική η καλύτερη λύση θα ήταν να λυθεί άπαξ και διαπαντό για όλε τι ευρωπαϊκέ γλώσσε σε όλε τι χώρε μέλη. Και έχω και κάτι άλλο να σα πω. Θα θέλαμε να δούμε, βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την ε, αναφορά, αλλά εμεί θα προτείνουμε να συζητηθεί το θέμα και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο πρόταση. Η δε πρόταση θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλες τις χώρες μέλη. Διότι όλοι θέλουν τα παιδιά τους να ομιλούν την μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστώ. Σφέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μίλαν Σβέρ, Σλοβαίνος. Ε, βέβαια, τα σλοβενικά ομιλούνται μόνο από δύο εκατομμύρια ανθρώπου, παρόλο που είναι η ορότερη γλώσσα του κόσμου, κατά τη γνώμη μου. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε να συμμετάσχουμε στην συνάντησή σα. Όπω ε, είπαν και οι συνάδελφοί μου, είμαι υπέρ τη διατήρηση ανοιχτή τη αναφορά και ω μέλο τη Επιτροπή ε, Πολιτισμού και ε, Παιδεία υποστηρίζω και την ιδέα να κατατεθεί προφορική ερώτηση προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο για την εκμάθηση γλωσσών από τα παιδιά. Και ιδίω για παιδιά που η μητρική τους γλώσσα τη χάνει να είναι από τις μικρότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι ορισμένε ε, περιστάσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες. Γι' αυτό και υποστηρίζω και την ιδέα να συζητηθεί στην Ολομέλεια το θέμα αυτό ώστε να φανεί καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυφωνίας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σοϊντρόβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία που πήραν οι Βούλγαροι συνάδελφοι. Εγώ είμαι από την Τσεχική Δημοκρατία Προέρχομαι λοιπόν από εκεί και κατανοώ πολύ καλά τα προβλήματά σας και τον προβληματισμό σας και εγώ θα επιθυμούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να παρακολουθεί καλύτερα ε, τα θέματα της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης ε, του γλωσσικού επίπεδου <clears throat> και των μικρότερων γλωσσών που μιλούνται από λιγότερα ε, λιγότερους πολίτες. Ε, και χαίρομαι γιατί η Κομισιόν δήλωσε ότι ε, δείχνει ενδιαφέρον και ότι θέλει να βοηθήσει. Συμφωνώ λοιπόν με την προσωπική προφορική συγγνώμη ερώτηση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πούμε μάλλον ότι ε, είναι πλούτος ε, η πολυγλωσία. Είναι δικιά μας ευθύνη να πούμε ότι ε, η πολυγλωσία είναι πλούτος και είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη, μέλη έχουν και αυτά βέβαια τις δικές τους υποχρεώσεις, αλλά εμείς κυρίως θα πρέπει να είμαστε οι θεματοφύλακες αυτού του πλούτου. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος Μαρλένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι από τη Βουλγαρία. Αλλά έχω τη βοηθό μου που είναι από την Βουλγαρία. Είναι εξαιρετική χώρα. Εγώ δεν αναφέρομαι στην χώρα μου, στην γλώσσα μου σαν μια μικρή γλώσσα. Είναι μια μεγάλη γλώσσα που μιλιέται από λίγους ανθρώπους. Βεβαίως εγώ υποστηρίζω την πρωτοβουλία ε, να ε, προωθήσουμε το θέμα αυτό, γιατί η εκπαίδευση βεβαίως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά όταν μιλάμε για γλώσσες γίνεται πλέον ευρωπαϊκό ζήτημα. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα, να φτάσει ακόμα και στην Ολομέλεια η συζήτηση αυτή. Δεν πρέπει να, να υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των γλωσσών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Το δεύτερο είναι ότι προωθούμε την πολυγλωσία. Είναι ένα σταθερό μήνυμα ε, που προωθούμε. Αλλά όταν κάποιος ε, μετακινείται ε, σε μια άλλη χώρα, σιγά σιγά χάνει την κουλτούρα του, τον πολιτισμό του. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και βεβαίως το πρώτο στοιχείο είναι η γλώσσα. Γιατί εάν κάποιος πηγαίνει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάνει σιγά σιγά την μητρική του γλώσσα, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε, προχωρήσουμε το θέμα παραπέρα. Ευχαριστώ, Μαρλένα. Ο κύριος Δαμπάσκη. Δύσκολο είναι να πω το όνομά σας. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έχω δύσκολο όνομα, λέει ο κύριος Δαμπάσκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η γλώσσα αποτελεί τη μνήμη, αποτελεί την ταυτότητα, την ιστορία. Ένα άτομο άνδρας ή γυναίκα, στην ουσία κατανοεί τον εαυτό του μέσω της γλώσσας πρωτίστως. Η γλώσσα μας διαμορφώνει και γινόμαστε αυτό που είμαστε. Συμφωνώ απολύτως. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεγάλη γλώσσα, μικρή γλώσσα. Εάν κανείς γνωρίζει μία γλώσσα και μπορεί να γράψει σε αυτήν ένα ποίημα ή μία, ένα τραγούδι, μα τότε είναι μεγάλη γλώσσα. Εάν έχουν γραφτεί και πολλά χρόνια πριν... Ε, Ε, όταν έχουν γραφτεί ιστορικά βιβλία ε, σε αυτήν την γλώσσα, τότε είναι μεγάλη γλώσσα. Ε, η ιστορία αυτή, η συζήτηση ξεκίνησε ήδη από το 1867 στην Βενετία, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τότε ε, είχε αναφερθεί ότι η Αγία Γραφή ε, μπορεί να ε, γράφεται μονάχα σε τρεις γλώσσες, αλλά τότε εκείνο είπε ότι θα πρέπει να γραφτεί και να προωθηθεί σε όλες τις γλώσσες. Αυτό είναι το σωστό. Εμείς παραμένουμε Βούλγαροι, Σλοβάκοι, Φιλανδοί, Δανείς ή Τσέχοι, αλλά μιλάμε ο καθένας τη γλώσσα του. Έστω και αν εδώ συνεργαζόμαστε και επειδή είναι και τα γενέθλιά μου κάντε μου το δωράκι να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Α, πολύ ωραία τα είπατε και σας συγχαίρω. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας. Είσαστε τόσο νέος, πολλά επιτεύγματα σας ε, περιμένουν. Και σας ευχαριστούμε πολύ γιατί τα είπατε πολύ όμορφα και με μεγάλη συγκίνηση. Κυρία Μποσκόρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα ως Αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού πρέπει να πω ότι υποστηρίζω πλήρως την ιδέα ε, να φτάσει το θέμα στην Ολομέλεια. και να έχουμε εκεί μια συζήτηση και επομένως να ε, ε, φέρουμε το θέμα σε υψηλότερο ε, επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό. Το θέμα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διασυνδεθεί ε, ή μάλλον να αναφερθεί στην προφορική ερώτηση ε, και να αναφερθεί και η πολυγλωσία και να ζητήσουμε ε, απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 15 εκατομμύρια ε, σε ολόκληρο τον κόσμο ε, μιλούν την ουγγρική γλώσσα. Έστω και αν μόνο 10 εκατομμύρια ε, ζουν στην Ουγγαρία, έχουμε μια διασπορά 5 εκατομμυρίων Ούγγρων σε ολόκληρο τον κόσμο και εμείς αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια για τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στη Σλοβακία, στην Κροατία, στην Ουκρανία, στην Σερβία, στη Σλοβακία έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, να μην χάσουν τον πολιτισμό τους και να μην αφομοιωθούν αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρίως γιατί προέρχεστε ε, από την Επιτροπή Πολιτισμού και είσαστε και αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγγελίεβα από την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία της Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, κυρία Κονεκτσίεβα, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια ε, για την μεγάλη της φιλοδοξία αλλά ε, και για την υποστήριξη και επιμονή που έδειξε και η ίδια καθώς και άλλες ε, οργανώσεις ε, του εξωτερικού. Η ιδέα είναι πάρα πολύ θετική. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τη γλώσσα σήμερα κυρίως, που, σε αυτή την περίοδο δηλαδή κυρίως, που η Βουλγαρία ε, κατέχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανέλαβε ε, πριν από ε, λίγο καιρό. Τον Δεκέμβριο ήδη είχαμε αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια συμπεριληπτική πραγματικά κοινωνία ε, επομένως, ε, ε, η Βουλγαρική Προεδρία προτίθεται να εργαστεί όσον αφορά το θέμα των βασικών προσόντων, key competencies. που περιλαμβάνουν και την ε, γλώσσα. Υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις ε, όπου δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι όσον αφορά το θέμα των, κεντρικών προσόντων, όλες οι χώρες δούλεψαν σκληρά και έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα των βασικών δεξιοτήτων εντός του εκπαιδευτικού ε, συστήματος και βεβαίως ε, μία από τις ε, κεντρικές δεξιότητες είναι η μελέτη και της μητρικής γλώσσας αλλά και ξένων γλωσσών. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα πολύ ωραία και σημαντικά ακούσαμε ήδη αλλά πραγματικά πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Η κυρία Κονακτσίεβα ζήτησε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός από όλα τα κράτη-μέλη που θα αναλάβει ε, την διενέργεια τελικών ε, εξετάσεων. Χαίρομαι γιατί ο κύριος ε, Μαλίνοφ επίσης αναφέρθηκε ε, στο θέμα αυτό και ενστερνίστηκε αυτήν την φιλόδοξη πρόταση. Ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από κοινού νομίζω ότι μπορούν να προωθήσουν το πλήρες ε, δυναμικό της εκπαίδευσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία και όπου το κάθε μέλος της κοινωνίας θα αισθάνεται καλά ενταγμένο στην κοινωνία αυτή, ότι ανήκει δηλαδή στην κοινωνία αυτή. Είναι σημαντικό οι πολίτες μας ε, να κατανοήσουν πλήρως, να συνειδητοποιήσουν την δύναμη της της ευρωπαϊκής ε, ε, ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και να προωθήσουμε και την θετική ανταγωνιστικότητα. Ε, τα βουλγαρικά ε, χρησιμοποιούνται και από 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο ε, τον κόσμο και επομένως ε, μπορεί μέσω της πρόθεσης και της γλώσσας να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν περισσότερες εταιρείες και στην Ευρώπη. Είναι ανοιχτή λοιπόν η Βουλγαρική Προεδρία για όλα. Θα πω τώρα κάτι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Βλαγκοντάρια που θα πει σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να τι αφιερώσουμε. Δυστυχώ δεν έχουμε. Ευχαριστούμε την αναφερομένη που ε, ήταν ε, σήμερα κοντά μας. Έχουμε ζητήσει και γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία δεν έχουμε λάβει ακόμη, να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, νομίζω, και αν συμφωνούν οι συναδελφοί μου, να ζητήσουμε ξανά την συνεργασία της Επιτροπής Πολιτισμού, να τους εξηγήσουμε τι λέχθηκε σήμερα στη συζήτηση. Ακούσαμε άλλωστε ότι θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω δράση, να αναλάβουμε περαιτέρω δράση, ίσως μια προφορική ερώτηση μαζί με μια νομοθετική επιτροπή, η οποία θα ήταν στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι καλός ο τρόπος αυτός για να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για το θέμα, ρωτώ εάν με υποστηρίζουν οι συνάδελφοι ώστε από πλευρά γραμματεία να ζητήσουμε τη συνεργασία τη Επιτροπή Πολιτισμού και μάλιστα έχουμε και τη μεγάλη τύχη να έχουμε κοντά μα τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτισμού. Λοιπόν, να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σα, Επιτροπή Πολιτισμού μαζί οι δύο επιτροπές μπορούμε να το προωθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Θα ήθελα επίσης να στραφώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την ευχαριστήσω για την πολύ περιεκτική παρέμβασή της. Σας ενθαρρύνω να σημειώσετε τα όσα λέχθηκαν σήμερα εδώ πριν από την επι... ενημέρωση για τις αρμοδιότητες για την διαβίου εκπαίδευση. Να εμπνευτείτε λοιπόν από την ανταλλαγή απόψεων που έγινε σήμερα και πολύ ευχαρίστω να επανέλθετε και να μα υποβάλλετε προτάσει για ουσιώδη βήματα προ τα εμπρό. Προ την αναφερομένη πάλι λέγω σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που θέσατε υπόψη μα την αναφορά σα. Η μητρική γλώσσα, οφείλω να τονίσω και πάλι, είναι η γλώσσα με την οποία εκφράζουμε τα όνειρά μα, τα αισθήματά μα, είναι η γλώσσα ακόμη και τη σιωπή. Και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Ότι χωρί τη μητρική γλώσσα, κοιτάξτε, η μητρική γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλε και όλου μα για να λειτουργήσουμε και στην επαγγελματική ζωή και στην ε, ε, προσωπική ζωή. Γι' αυτό να σημειώσουμε την σημασία όλων των ε, ε μητρικών γλωσσών. Είμαστε, όπω γνωρίζουμε, ενωμένοι στην πολυφωνία. Ευχαριστώ και όλους τους Βουλγάρους συναδέλφους και θεωρώ ότι με την σιωπή σας με υποστηρίζετε. Προχωρούμε για τον κύριο Ζαμπάσκι. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Παρακαλώ, όσοι και όσες επιθυμείτε να ε, αποχωρήσετε, σας παρακαλώ το της ήχος, διότι εδώ συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Η κυρία Μίτση, Προεδρεύουσα, αρχίζουμε τώρα με... Αρχίσαμε... Ή ε, μάλλον, δεν έχει έρθει ακόμα ο αναφερόμενος ή αναφερομένη της αναφοράς για το σημείο 9. Είναι παρούσα ή παρόν? Άρα δεν ήσασταν πριν εδώ, είστε εδώ τώρα. Μάλιστα. Ε, πρόκειται για την 0954-2017 σχετικά με εικαζόμενη μη τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας από το γερμανικό κράτος. Έχετε το λόγο κυρία. Μάλιστα, με ακούτε. Ωραία. Πρόκειται για το άρθρο 9 παράγραφος 3 Ευρωπαϊκού Κανονισμού του 2006 όπου περιλαμβάνεται ο όρος χρόνος εργασίας. Πρέπει όμως να λέει χρόνος οδήγησης και εργασίας, ώστε οι οδηγοί να ε, ε, γράφουν στον ε, ταχογράφο όλες τις ώρες εργασίας. Στην υπόθεση Κέρτς, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημειώνει ότι η ώρα εργασίας των οδηγών αρχίζει από το κέντρο το κέντρο διαβίωση, δηλαδή από το σπίτι τους. Τους στέλνουν να πάρουν το φορτηγό και ξεκινούν μετά από αυτό, ξεκινά δηλαδή η βαρδιά τους και φτάνουν να είναι ξύπνοι 30 ώρες. Και πώς θα ανταποκριθούν στα καθήκοντα του επαγγελματό τους να μείνουν ξύπνοι τόσες πολλές ώρες. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Και δεν είναι δυνατόν και από την άποψη οδική ασφάλεια, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, λέει εκεί ώρες οδήγησης και ώρες εργασίας. Πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ώρα εργασία, ώστε κάθε αστυνομικός, κάθε επιθεωρητής να μπορεί να εξετάζει αυτός ο οδηγός πόση ώρα, πόσες ώρες βρίσκεται στον ε, αυτοκινητόδρομο. Τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο άνθρωπο αυτός είναι ικανό ακόμη να οδηγήσει. Τι μπορούμε να αναμένουμε από αυτόν. Μπορεί να οδηγήσει το μεγάλο αυτό όχημα στους αυτοκινητοδρόμους. Ήθελε να συμπληρώσει κάτι ο ε, κύριος που κάθεται εξ αριστερών Να συμπληρώσω επ' αυτού ότι η έδρα του φορτηγού αυτοκινήτου μέσα στην παγκοσμιοποίηση δεν συμπίπτει με την έδρα της επιχείρησης. Η έδρα του φορτηγού από την έδρα της επιχείρησης συχνά είναι διαφορετικές. Υπάρχουν πολλές εταιρείε εικονικές, οι οποίες παρκάρουν τα φορτηγά αυτοκίνητα σε κάποιο χώρο στάθμευσης που δεν έχει καμία σχέση με την έδρα τους. Ο οδηγός του αυτοκινήτου λοιπόν σήμερα για τις ε, μεταφορές εξωτερικού πρέπει να μετακινηθεί προς το φορτηγό αυτοκίνητο από κάπου, οπουδήποτε, στην Ευρώπη, στη Γερμανία και τότε αρχίζει η, δεκα, η δεκάωρη βάρδιά του. Επομένως, η συνολική ε, διάρκεια που περιλαμβάνεται στο 9 παράγραφος 3 του 561.06 είναι, αναφέρονται εκεί ως άλλες εργασίες, το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οι ώρες εργασίας μπορεί να είναι η ε, διαθεσιμότητα για να είναι δηλαδή έτοιμος να εργαστεί. Ώρες οι οποίες δεν καταγράφονται στον ψηφιακό ταχογράφο. Πρόκειται για διακινδύνευση. Θα πρέπει μόνο να λέει ώρα οδήγησης και εργασίας, αντί να λέει για άρες δραστηριότητες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσφαλμένα το περιλαμβάνει στις κατευθύνες γραμμές της. Είναι απολύτως εσφαλμένο και πρέπει να διορθωθεί. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα κυρία Μίτση. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ ε, να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού καλωσορίσω τους δύο αναφερομένους. Η νομοθεσία για, το κανονισμό 561 του 06 απαιτεί ο οδηγός να καταγράφει κάθε εργασία εκτός οδηγήσεως είτε με άλλο εργοδότη είτε με τον ίδιο εργοδότη εντός ή εκτός ε, τομέως μεταφορών, να τα καταγράφει στον ταχογράφο. Αυτά τα απαιτεί ο κανονισμός. Υπάρχουν και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του κανονισμού που ορίζουν ότι ο οδηγός καταγράφει και την διάρκεια μετάβασης για να λάβει το φορτηγό το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, δηλαδή για φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων μεικτού βάρου. Όταν λοιπόν μεταβαίνει στο φορτηγό αυτοκίνητο για να το αναλάβει, αλλά και για την επιστροφή του από την τοποθεσία του φορτηγού αυτοκίνητου. Αυτά πρέπει να καταγράφονται με το χέρι στον ταχογράφο όταν αναλαμβάνει για πρώτη φορά την οδήγηση του φορτηγού αυτοκινήτου των 3,5 τόνων. Αυτά απαιτούνται ήδη από το κείμενο του κανονισμού. Υπάρχουν βέβαια διαφορές δεν ξέρω αν θέλετε να μπω στις διαφορές τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς καταγράφονται τα στοιχεία αυτά. Αν όμως ένας οδηγός οδηγεί το φορτηγό άνω των 3,5 τόνων προς τον τόπο όπου θα φορτωθεί, αυτό είναι driving time. Εάν το φορτηγό εκπίπτει το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, τότε αυτό θεωρείται άλλες εργασίες. Εάν πάρει το τρένο ή αν ταξιδεύσει μαζί με κάποιον άλλο, αν την οδηγεί ο ίδιος δηλαδή ο οδηγό και δεν έχει πρόσβαση σε κουσέτα για να ξαπλώσει, αυτό μπορεί να θεωρηθεί άλλη εργασία ή μπορεί να θεωρηθεί περίοδος διαθεσιμότητας. Αυτά για το τεχνικό τμήμα. Έχουμε επίσης και την οδηγία, οδηγία 2002-15, που ορίζει τα ανώτατα όρια της εργασίας. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο τον κανονισμό αλλά έχουμε και την οδηγία χρόνου οδηγήσεως ή χρόνου εργασίας που λαμβάνει υπόψη τον χρόνο οδηγήσεως, άλλες εργασίες και περιόδους διαθεσιμότητας. Και που ξεκαθαρίζει επίσης ότι ο οδηγός δεν θα πρέπει να εργάζεται περισσότερο κατά μέσον όρο από 48 ώρες την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να παρατηραθεί σε 60 ώρες την εβδομάδα μόνο εάν μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών δεν ξεπερνά το μέσον όρο των 45 ώρων την εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν την ομοθεσία αυτή που περιορίζει τον χρόνο οδηγήσεως όπως και τον χρόνο εργασίας. Ε, αυτό που μπορώ να προσθέσω ακόμη είναι ότι βρισκόμαστε στη φάση αναθεωρήσεως του 561 κανονισμού μέσα στα πλαίσια του πακέτου μέτρων κινητικότητας από τον Μάιο του 2017 και τώρα βρίσκεται στη φάση της διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αυτό που εξετάζουμε είναι να βελτιώσουμε την συμμόρφωση των χωρών μελών για τον έλεγχο των ανώτατων ορίων εργασίας και περιλαμβάνουμε και τις εικονικές εταιρείες, δηλαδή αυτές τις εταιρείες γραμματοκιβωτίου. Θέλω να προσθέσω ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αναδιετία δεδομένα από τις χώρες μέλη σχετικά με το πώς ελέγχουν την εφαρμογή του 561 για, την, ε, για τον χρόνο εργασίας και η Γερμανία τα πηγαίνει θαυμάσια. Κάνει τους καλύτερους ελέγχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνουμε και ποιοτικά δεδομένα από τις χώρες μέλη για την οδηγία χρόνου εργασίας. Με τις προτάσεις που ανέφερα προηγουμένως αποσκοπούμε στο να λάβουμε και ποσοτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης με την οδηγία χρόνου εργασίας. Θεωρούμε ότι οι ανησυχίες των αναφερομένων αντιμετωπίζονται ήδη και ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και με, την, ε, με τους εργασίας είτε ήδη από την νομοθεσία είτε πρόκειται να αντιμετωπιστούν στην αναθεώρηση της ε, σχετικής νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος κυρία Βίξτρον που επανέκαμψε. Ευχαριστώ την Μαρλένε που με βοήθησε. Χρειάστηκε να πω για λίγο. Και τώρα βεβαίως το λόγο έχετε εσείς, Πέτερ Γιάρ. Και ο Γιάρος Λαβαλένσα που επεξεργάστηκε την αναφορά είπε κάποια πράγματα να πω. Ευχαριστώ πρώτα για την αναφορά, ευχαριστώ τους αναφερομένους. Και αν κατάλαβα καλά, πρόκειται εδώ για ένα κενό ρύθμισης. Ομολογώ ότι δεν είμαι εμπειρογνώμων για θέματα μεταφορών. Ίσως με κάποιο σύντομο τρόπο ε, πρόκειται για το φορτηγό, μέσα στο φορτηγό. Λειτουργεί λίγο πολύ η νομοθεσία, υπάρχουν δηλαδή ώρες ανάπαυσης, ώρες οδήγησης και ούτω καθεξής. Ή αμφιβολίες των αναφερομένων, ίσως πρέπει κανείς να αποστασιοποιηθεί από μια ρομαντική εικόνα του επαγγέλματος του φορτηγού, ότι δηλαδή ο οδηγός παίρνει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, κάνει μια διαδρομή 10 λεπτών και ανεβαίνει στο φορτηγό του αυτοκίνητο. Αυτά τα πράγματα είναι πιθανόν να μην υπάρχουν πια. Πηγαίνει, για μεγάλο χρονικό διάστημα μπαίνει στο φορτηγό και δεν ξανακατεβαίνει. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ρυθμίσει, γιατί αν δεν υπάρχουν ρυθμίσει, λείπει και η ασφάλεια δικαίου. Αν ρωτήσετε ένα φορτηγό αυτοκινήτου θα σα πει «Α, είμαι ξεκούραστος» και μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο. Τώρα, μιλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άνω των 3,5 τόνων. Είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται ρύθμιση την οποία συντάσσει τώρα αναθεώρηση. Νομίζω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά εφόσον βρίσκεται σε προπαρασκευή αναθεώρηση νομοθεσίας να τα διαβιβάσουμε αυτά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία θα χαρεί να λάβει και κάποιες επισημάνσεις από την ίδια την πράξη, από την πρακτική σκοπιά δηλαδή του, της ρύθμισης και του επαγγέλματος. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών, να παρακαλέσουμε να γνωμοδοτήσει και τα αιτήματα των αναφερομένων να τα περιλάβει στη νέα νομοθεσία που θα προτείνει. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος κυρία Κρότσα. Η κυρία Πρόης, ως μέλλον της Επιτροπής Μεταφορών έχω να σας πω ότι χθες διεξήχθη η πρώτη ακρόαση και η σκιώδης η μας τόνισε ακριβώς τα θέματα αυτά. Δηλαδή βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Βεβαίως και σημειώνω τις ε, προτάσεις των αναφερομένων, μιας και είμαι και συντονίστρια κιόλας, θα εξετάσω με μεγάλη προσοχή την αναφορά και θα παρακολουθήσω κατά πόσο η κίνηση γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κράους, παρακαλώ, αναφερομένη, να λάβει πάλι το λόγο. Ε, ε, ε, Αν με επιτρέπετε να απαντήσω εγώ, λέει ο αναφερόμενος, είχα πει στην αρχή ότι η έδρα του φορτηγού και η έδρα της επιχειρήσεως διαφέρουν, ιδίως στο ανατολικό της Ευρώπης δεν συμφωνούν. Οι έδρες των εταιριών και οι έδρες των φορτηγών αυτοκινήτων απέχουν καμιά φορά 50, από 50 έως 1000 χιλιόμετρα οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Δεν συμπίπτουν πλέον. Παλαιότερα η έδρα της ε, επιχειρήσεως ίσως ήταν 20-30 χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο στάθμευσης του φορτηγού αυτοκινήτου. Σήμερα όμως χρειάζεται να κινηθούν οι οδηγοί από το σπίτι τους, από το σπίτι τους σημειώνω, με ιδιωτικά αυτοκίνητα εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αυτά πρέπει να θεωρηθούν χρόνος οδήγησης και εργασίας. Είτε είναι 50 χιλιόμετρα είτε είναι 1000 χιλιόμετρα. Πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και αυτά πρέπει να θεωρηθούν χρόνος εργασίας. Αυτό που λέει το 9-3 άλλες εργασίες πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να λέει χρόνος οδήγησης και εργασίας. Και με τον τρόπο αυτό λύνεται το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δυο σας που ήρθατε σήμερα να μας τα πείτε. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση αυτή. Είπαμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά και είναι καλή ιδέα πράγματι να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Μεταφορών για να γνωμοδοτήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, βεβαίω όλες και όλους. Καλή επάνωδο ε, στα σπίτια σας και ελπίζω να σας φάνηκε καρποφόρα η επίσκεψή σας στις Βρυξέλλες. Ας ε, επιστρέψουμε τώρα στην ε, αναφορά υπαριθμών, μάλλον στο θέμα υπαριθμών 11, Πρόκειται για την 0907 του 2009. Είναι ε, παρόντες οι αναφερόμενοι. Πρόκειται για το κλουμπ Ντεντονιάνα σχετικά με την επιδείνωση των συνθήκων στο Εθνικό Πάρκο Δονιάνα. Πρόκειται για τον κύριο Γκονζάλες και ενδεχομένως τον κύριο Καναδάς και τον κύριο Καζανόβα. Η Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε συντομότατοι γιατί μας μένουν μόνο 20 λεπτά για να συζητηθεί το θέμα σας. Ορίστε. Καλό μεσημέρι. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον Ιούνιο του 2013, όπου ήδη με την παρουσία μας σε τούτη την Επιτροπή Αναφορών ε, ε, ε, ήρθαμε για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και υποβάλαμε το θέμα μας και θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την Επιτροπή σας εδώ ακριβώς ε, για την ευαισθησία που έδειξαν όσον αφορά το θέμα του, που μας απασχολεί. Ε, είναι χιλιάδες οι πολίτες που στην Ισπανία και στην Ευρώπη αναρωτιούνται η δομάνια, ε, η δωνιάνα συγγνώμη, είναι πολιτιστική κληρονομιά, ε, είναι ε, καταφύγιο βιοσφαίρας, είναι ακριβώς το κατάλληλο σημείο έτσι ώστε να εξορυχθούν 860.000 τετραγωνικά κυβικά μέτρα αερίου ε, σε αυτήν την ερώτηση αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ε, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να δίνεται έγκριση για έργα που περιλαμβάνουν εξόρυξη και αποθήκευση και μεταφορά φυσικού αερίου ε, σε αυτό το σύμβολο της φυσικής ποικιλομορφίας ήδη από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πολλές φορές ήρθαμε σε επαφή και παρουσιαστήκαμε είτε εις διάφορα φόρα είτε ακριβώς ακριβώς εις τον διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας. Επίσης ήρθαμε σε επαφή ε, με ε, εμπειρογνώμονες καθώς επίσης ε, και με το Γεωλογικό και Εξορυκτικό Ινστιτούτο της Ισπανίας. Όλοι συμφωνούν ότι η τοποθεσία δεν είναι η κατάλληλη λόγω ακριβώς της περιπλοκότητας του γεωδυναμικού μοντέλου της περιοχής. Επίσης γιατί δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα. Ε, οι μελέτες περιβαλλοντικής επιπτώσεως ε, δεν περιέλαβαν ποτέ ανάλυση όσον αφορά ε, την συνολική επίπτωση των τεσσάρων σχεδίων που αφορούν το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους μεμονωμένα έργα στην να Θα πρέπει να μετρηθεί ο συλλογικός τους αντίκτυπος ε, μας λένε στην αρχή να τα κάνετε, να ξεκινήσουν τα έργα και μετά θα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ναι, αλλά τότε οι επιπτώσεις ε, δεν θα μπορούν να αντιστραφούν. Ε, τον προηγούμενο ε, Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει μία μελέτη την οποία απέκρυψε η κυβέρνηση όπου αναφέρεται ότι αυτό το, το πρόγραμμα του φυσικού αερίου μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς ε, κινδύνους. Ε, θα πρέπει εδώ επομένως ε, να εφαρμοστεί η αρχή της πρόληψης, έτσι όπως αναφέρεται και στο άρθρο 191 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 2 του Ισπανικού Νόμου 21-2013 για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και του άρθρου 2G του νόμου 42-2007 της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιοπικιλότητας. Ακριβώς δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά την Δονιάνα. Εμείς αισθανόμαστε ότι ε, οι κάτοικοι της Ανταλουσία, ε, της Ισπανίας αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκονται κοντά μας όταν ζητάμε την προστασία της Επιτροπής Αναφορών ενώπιον των πράξεων της κυβέρνησης της Ισπανίας σε σχέση με αυτό το project. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Επιτροπή Αναφορών να απευθυνθεί στην κυβέρνηση της Ισπανίας, να ζητήσει να σταματήσει άμεσα ε, το ε, project μαρίζμα Occidental, το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει να εκτελείται. Δεύτερον, να ζητήσουμε την συνολική ε, αντιμετώπιση και αξιολόγηση των τεσσάρων προγραμμάτων στα οποία με τρόπο απατηλό έχει μοιραστεί το κεντρικό project και που δημιουργεί πρόβλημα εις τον υδροφόρο ορίζοντα 27 της Ντονιάνα. Τέλος, ζητούμε ε, να οργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτόπου διαρευνητική αποστολή έτσι ώστε να δει και η διεισόμαση ε, τα προβλήματα και τους κινδύνους αυτού του προγράμματος. Και εσείς εδώ ε, έχετε ιστορική ευθύνη να σώσετε έναν μοναδικό φυσικό τόπο όπως είναι αυτός της Δονιάνα η συντήρηση του οποίου μπορεί πραγματικά ε, να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι εγωιστικά και καταχρηστικά ε, μπορούν να προκαλέσουν ανεπίστρεπτα προβλήματα ε, και εάν σώσετε την Τονιάνα οι μελλοντικέ γενιές θα σας ευγνωμονούν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια εξαιρετικά σύντομη απάντηση αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε λέει ο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται ε, την άποψη των ε, αναφερομένων, ε, μάλλον τον προβληματισμό των αναφερομένων για την Δονιάνα και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ, διότι η Δονιάνα είναι προστατευόμενο εθνικό πάρκο και επίσης και έχει πολλές προστατευόμενες περιοχές από το δίκτυο Natura 2000. Κατά την έννοια αυτή η πρώτη αναφορά αυτού του συνόλου αναφέρεται στην επιδίνωση των συνθήκων ε, των διατημάτων στο Εθνικό Πάρκο της Δονιάνα. Επίσης ε, γίνεται λόγος ε, για το πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα και των ε, ε, αποθηκών ε, των ταμιευτήρων μάλλον υδάτων που είναι απαραίτητη για την προστασία του δικτύου Natura 2000 και της βιοπικιλότητας. Εδώ έχουμε την οδηγία για τα ύδατα, καθώς επίσης και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, καθώς επίσης και την οδηγία για τα ενδιατήματα. Ναι, ε, είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε λάβει πάρα πολλά στοιχεία και από τις Ισπανικές αρχές αλλά και από τους αναφερόμενους. Όσον αφορά ε, τα, τις εργασίες εξόρυξης και αποθήκευσης ε, φυσικού αερίου, που αποτελεί θέμα επίσης της αναφοράς, έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τις αιτιάσεις που αναφέρονται, έχει ξεκινήσει, λέω, διερευνητική ε, διαδικασία. Αυτή η διερεύνηση ως ήθιστε αφορά την σωστή εφαρμογή ε, της ε, ισχύουσας νομοθεσίας από πλευράς των Ισπανικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά από τη διερεύνηση του θέματος είναι ότι πράγματι πρόκειται για τέσσερα project τα οποία έχουν υποβληθεί σε διαφορετικές διαδικασίες ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου από πλευράς νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί παράβαση. Διότι αυτό που απαιτεί η νομοθεσία είναι να ληφθούν υπόψη όλα τα όλες οι σορευτικές επιπτώσεις οι οποίες μπορούν ε, να προκύψουν και επομένως να γίνει και συνολική αξιολόγηση των ε, projects αυτών. Η Κομισιόν έχει επίσης λάβει πληροφορίες ε, ότι ε, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αυτές με ε, θετική έκβαση όσον αφορά την τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ε, η Κομισιόν αξιολόγησε την μελέτησε την αρνητική αξιολόγηση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν τόσο από πλευράς των αναφερομένων όσο και από πλευράς κάποιων οργανισμών και ε, ζητήθηκαν κάποιες ε, ε, διορθώσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην οδηγία και που παραπέμπουν σε τα δικαστικά ένδικα συγγνώμη, μέσα των κρατών μελών. Λάβαμε επίσης ε, πληροφορία, την πληροφορία ότι η Ανδαλουσία έχει ξεκινήσει διαδικασία διοικητικής προσφυγής ε, για αυτά τα τέσσερα projects. Η Κομισιόν σε αυτές τις περιπτώσεις ε, ως ήθιστε δεν κάνει παράλληλες διερευνήσεις ε, και ε, από τη στιγμή που βρίσκεται ενώπιον του δικαστού το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον ε, του Εθνικού Δικαστού και μετά. Ευχαριστώ πολύ η Κομισιόν αναφέρθηκε στην Ανδαλουσία. Έχουμε εδώ τον Ανδαλουσιανό διαμεσολαβητή. Για πολύ λίγο θα σας δώσω το, το λόγο. Βρίσκομαι ενώπιον σας ε, διότι ε, αναφέρομαι ε, σε αυτήν την πρόσκληση της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου σας για να αναφερθώ για ένα θέμα, σε ένα θέμα το οποίο μας επηρεάζει όλους. Την διατήρηση των ευνοϊκών συνδικών στο Εθνικό Πάρκο Δονιάνα που μπορούν να επιδεινωθούν από το, τις εργασίες εξόριξης και μεταφοράς φυσικού αερίου. Το θέμα αυτό προβληματίζει τους πολίτες ε, αλλά και πολλά μέλη ε, της ε, επιστημονικής κοινότητας. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι με τις πληροφορίες που σας έχουμε περιλάβει και στα έγγραφα και στο φάκελο που σας έχουμε υποβάλει, ε, το, τα project στην Δονιάνα δεν συνάδουν με την αρχή ε, της ε, πρόληψης και της σωστής συντήρησης του Εθνικού Πάρκου της Δονιάνα. Εξηγούμε και αιτιολογώ. Πρώτον, δεν εφαρμόστηκε η κοινοτική οδηγία η ε, οι ε, περιβαλλοντικές αρχές της Ανδαλουσίας ε, οι αρχές του συνηγόρου του πολίτη της Ανδαλουσίας η αξιολόγηση της επιστημονικής κοινότητας της Ανδαλουσίας που ζήτησαν κοινή αξιολόγηση των τεσσάρων τμήματων του προγράμματος του project αυτού. Θα πρέπει από κοινού να μελετηθούν τα τέσσερα ε, επιμέρους project έστει ώστε να αξιολογηθεί ο σορευτικός αντίκτυπος. Δεύτερον, έτσι όπως ε, ε, προβλέπεται ε, και από τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου των τεσσάρων τμήματων δεν υπάρχει ταυτοποίηση ε, των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από την έγχυση φυσικού αερίου στο υπέδαφος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί και το στοιχείο αυτό στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου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 Επίσης δεν είναι ε, δυνατόν να μην ε, ε, βρούμε παράλληλα στοιχεία με την πάυση της πλατφόρμας Καστόρ που αφορούσε ακριβώς και την εξόριξη φυσικού αερίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ισπανίας, ο Εισαγγελέας της Ανδαλουσίας αναφέρουν ότι υπάρχει, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και ικανή αμφιβολία ε, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα projects αυτά. Το γεωδυναμικό μοντέλο της περιοχής είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Έχετε ήδη φτάσει στα τρία λεπτά όμως. Δεν θα έχουμε διαρμηνία σε λίγα δευτερόλεπτα και έχω ακόμα τόσους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μας ε, είπατε όλα αυτά τα τόσο σημαντικά. Θα συνοψίσω λοιπόν, ε, οι συντονιστές ε, πήραν την απόφαση ότι θα σταθούμε στο πλευρό σας. Έχω την κυρία Καμπεσόν, τον κύριο Μιράντα. Αγγουιλέρα Γκράσια, Γκαρσία Ιστουγκάιζ, Μπενίτου, Λόπες, One minute each, starting with Soledad. Ένα λεπτό καθένα καθένας, Πολύ σύντομα, ναι, αφού μου δίνετε ένα λεπτό. Είμαι πολύ... με, με εντυπωσιάζει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι είχαμε κάνει μια άλλη αναφορά και με τον ίδιο λόγο, με το ίδια αίτια. Σήμερα είναι μια πρόκειται για παράβαση πλέον, αλλά με εντυπωσιάζει όχι μόνο γιατί δεν ε, έχετε δίκιο, αλλά γιατί υποχρεώνεται την περιφέρεια της Ανδαλουσίας ε, να πάει στα δικαστήρια. Δηλαδή να στείλετε μια επιστολή στην κυβέρνηση της ε, Ισπανίας ε, και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, παραβαίνετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τέλος. Τι υπάρχει που σας εμποδίζει να δράσετε και Εάν σταματήσει λοιπόν τελείως αυτό το, αυτός ο αγωγός, η κατασκευή αυτού του, του αγωγού, ε, ε, θα έπρεπε να γίνει από πλευρά σας. Γιατί μόνο η περιφέρεια της Ανδαλουσίας έχει κάνει κάτι για να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ευχαριστώ, Ζολεδάδη, κυρία Μιράντα. Αυτό το, αυτή η αναφορά είναι πολύ δίκη και μάλιστα οι ε, αναφέροντες ε, πέντε χρόνια ταλαιπωρούνται. Είναι κλασική περίπτωση. Το είδαμε και στο project Castor με τα γνωστά αποτελέσματα. Και η Κομισιόν δεν τρέπεται με αυτές τις δηλώσεις, γιατί πώς μπορεί να μας στέλνει κατευθείαν ε, στα δικαστήρια εφόσον υπάρχει υποστήριξη από τον διαμεσολαβητή και από την ε, τοπική διοίκηση. Αυτό εδώ και σήμερα ψηφίσαμε ότι θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία. Υπερψηφίσαμε εμείς αυτή την Επιτροπή. Και θέλω να θυμίσω ότι στη συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα εγκρίθηκε επίσκεψη στη Δονιάνα. Και εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. Ευχαριστώ. Μαρσελέση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα σας πω ότι, δεν, ότι με εντυπωσιάζει αυτή η απάντηση. Να μας στέλνετε στα δικαστήρια, όταν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει αρχίσει η διαδικασία κατά παράβαση έχετε, και λέτε εδώ στους ε, αναφέροντες να τρέξετε στα δικαστήρια, ενώ έχουμε συγκεκριμένη, εγκεκριμένη πολιτική στην Επιτροπή Αναφορών που λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά θα έπρεπε να έχετε δουλέψει νωρίτερα, να έχετε αντιδράσει νωρίτερα για να μην ε, ε, χάνετε την εικόνα εικόνα σας και να δίνετε τέτοια άσχημη εικόνα της Υπήρου μας. Εμείς δεν θέλουμε άλλο, άλλη υπόθεση καστορτίνη. Είχαμε μια φορά στην Ισπανία, δεν θέλουμε και δεύτερη τέτοια υπόθεση. Γι' αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει γιατί πρόκειται για κληρονομιά της ανθρωπότητας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή για αυτό το τόσο φυσικό δρυμός. Και έπειτα, χαίρομαι πολύ που αποφασίστηκε η επίσκεψη και που υπάρχει ένας ε, αναφέροντας εδώ που θέλει να μιλήσει, να δοφήσουμε άλλον ένα λεπτό, να μιλήσει γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι στην Ανταλουσία. Ναι, εγώ θέλω να σας δώσω για μια ώρα, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν θα έχουμε πια διερμηνία. Κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Αγγιλέρα Γκαρσία. Κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εμένα με εντυπωσίασε πώς απάντησε η ε, Κομισιόν και μάλιστα <coughs> ε, είναι κακό αυτό. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε η Σολεδάδη Καμπεσόν. Να πω και εγώ ότι η ε, Περιφέρεια τη Ανδαλουσία έχει στείλει επιστολή στην Επιτροπή μα και θέλω να το θυμίσω γιατί πιστεύω πω είναι πολύ σημαντικό. Η διοίκηση τι έκανε, να ανησυχεί και να ασχολείται με αυτό το θέμα που δημιουργεί η κρατική κυβέρνηση τη Ισπανία και μάλιστα θα ήθελα να λάβετε υπόψη επιπλέον ότι υπήρξε πρόσκληση της ε, Περιφέρειας Ανταλουσίας να επισκεφθείτε και να δείτε επιτόπια τι γίνεται. Νομίζω πως ε, πρόκειται για είναι πρόβλημα γενικής αξιολόγησης αυτού του project. Είναι πολύ βλαβερό για τον φυσικό δρυμό της Δονιάνα και η διοίκηση της Ανδαλουσίας λέει πως αυτή το project είναι ε, καταστροφικό για τη Δονιάνα που θα έπρεπε να προστατευτεί πάνω απ' όλα. Μάλιστα ο κύριος Τουρκάης, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ και, και το ε, ε, ε, θέλω να απαντήσω στον αναφέροντα ότι η κυβέρνηση πάντοτε εργάζεται προς το γενικό και συμφέρον όλων. Θέλουν να θεσπίσουν και κρατικούς και κοινοτικού νόμους. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θετικέ εκθέσεις που έγιναν και που έχουν γίνει στη διαδικασία αυτή από τη διοίκηση της Ανδαλουσίας, μάλιστα της Ανδαλουσίας και η κυβέρνηση Ανταλουσία έκανε ένα βήμα πίσω Εδώ. Εσείς αναφέρεστε σε μια ανέκθεση του Ισπανικού Ινστιτούτου Γεωλογίας και Εξόριξης που λέει και συνέλεξε συγκεκριμένα μέσο στις 16 Ιουλίου του 2016 και είπε ότι είναι μία μελέτη και ότι πρέπει να φτάσει στα δικαστήρια. Σας ευχαριστώ διακόπτη πρόεδρος. Διακόπτη η πρόεδρος του ομιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, λίγο έχετε ξεπεράσει τα όρια. Τώρα σας παρακαλώ. Εντάξει. Ο κύριος Μπενίτο, ναι, ναι, άμα τελειώσει ο χρόνος μας θα αφήσετε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα της Δονιάνα, αρκεί να το επισκεφθεί κανείς, όπως ήδη αποφασίστηκε σε αυτήν την Επιτροπή. Είναι ήδη σημαντικό αυτό να το επισκεφθείτε για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χώρος. Είναι ο χώρος ε, ε, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, όχι μόνο ε, επειδή είναι τόσο παλιός, αλλά και λόγω της σημασίας της φυσικής. Είναι ένας φυσικός δρυμός ε, που είναι κλειδί Ε, για την ανάπτυξη. Δεν, δεν πρέπει λοιπόν να επιτραπεί αυτό το έργο το οποίο θα έχει, α, πρόσλε, ε, θα έχει πολύ σημαντικές βλαμπερές συνέπειες. Η αρχή της προφύλαξης δεν λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρνηση της Ισπανίας, θέλει να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καλά θα έκανε να ε, επιμείνει σε αυτό και να κρατήσει σαφή θέση ενώπιον αυτού του κινδύνου που θα γίνει σε τέτοιο τόσο σημαντικό δρυμό. Ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Λόπες Βερεμέχο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να πω, να τονίσω τα εξής. Πρώτον, καταρχάς στηρίζω τους αναφέροντες και τις διεκδικήσεις τους που είναι μάλιστα ε, και ξεκάθαρα, ξεκάθαρες και ε, πολύ τεκμηριωμένες. Ε, και με το παραπάνω. Έπειτα να πω ότι όντως εδώ πρόκειται για την προδοσή... Ε, ε, ήρθε μια επιχείρηση να κάνει ένα κερδοσκοπικό project ε, αντίθετο προς το γενικό συμφέρον και προς το συμφέρον του ίδιου μας του, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναν φυσικό δρυμό που προστατεύεται όπως είναι ο φυσικός δρυμός της Δονιάνα. Μην μου λέτε πως δεν υπάρχουν κομματικά συμφέροντα. Υπάρχουν και εδώ έχουν υποστηριχθεί από την εταιρεία η οποία στηρίζει αυτό το κερδοσκοπικό σχέδιο, project. Η διοίκηση της Ανδαλουσίας έχει κάνει τέτοιες ε, εκτιμήσεις και χάρη στην κοινωνική πίεση και η Κομισιόν να σταματήσει τις δικαιολογίες ε, και άμεσα να σταματήσει αυτό το έργο και να απαιτήσει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί κανόνες. Αυτό οφείλει να κάνει αυτός ο θεσμός. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χέμερσταϊν Καζανόβα για ένα λεπτό, γιατί οι διερμηνείς μας έδωσαν έναν ε, ε, λίγο χρόνο παραπάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι εδώ εξ ονόματος του Αουρέλιο Κονθάλες Πόσα. Από την ε, Ένωση Δηλαδή, ε, ήμασταν εδώ και το 2013 σε σχέση με τις διεκδικήσεις που γίνονται εκεί ε, λόγω της κερδοσκοπικής επιχείρησης ε, είναι τρεις. Ε, τρεις οι εταιρείε που θέλουν να εκμεταλλευτούν εκεί την περιοχή ε, παραβαίνοντας κάθε κοινοτική νομοθεσία. Να σας πω ότι εσείς θα πρέπει να σταματήσετε αυτούς τους απάνθρωπους και τα project αποθήκευσης της γκάς και η, εξαγω... να, να γίνει πραγματικότητα. Να το απαγορέψετε αυτό. Εμείς ανέκαθεν υποστηρίζαμε ότι οι βιομηχανικές εργασίες που κάνουν αυτές οι τρεις επιχειρήσεις μέσα στο φυσικό δρυμό της Δονιάνα δεν τηρούν καμία νομοθεσία και κανένας δεν ήρθε να τις αξιολογήσει από κοινού. Γι' αυτό καταγγέλουμε εδώ ότι οι ισπανικές αρχές είναι συνένοχες στη μετατροπή και στην ε, καταστροφή του φυσικού πάρκου της ε, Δονιάνα και της μετατροπής τους σε μία, ένα χημικό ε, κέντρο της Ουέλβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαρίστω σας ανακοινώνω ότι σήμερα οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια ε, επίσκεψη εξεταστική των πραγμάτων, ειδικά στην περιοχή σας, για το δεύτερο εξάμεινο του φετινού χρόνου. Νομίζω θα είναι πολύ επίκαιρη η επίσκεψη αυτή. Θα εξετάσουμε τις διάφορες πλευρές, διάφορες πτυχές του θέματος και θα επανέλθουμε σε εσά του αναφερομένου και θα έρθουμε να σα δούμε στην περιοχή σα. Θα ξαναειδωθούμε δηλαδή, δεν θα χρειαστεί όμω να ταξιδεύσετε εσεί, θα έρθουμε εμεί να σα δούμε. Τώρα, για το λόγο αυτό, είναι τιμή για μένα να πω ότι διατηρούμε τις αναφορές ανοιχτές, ζητούμε περαιτέρω εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα γραπτός, ώστε να συμπληρώσει τα όσα είπε και προφορικός. Θα στείλουμε και επιστολή στην Χούντα Ανταλουσία που θα ζητούμε να εξηγήσουν τα μέτρα που λαμβάνουν και θα εκφράσουμε και τις ανησυχίες μας για την επιδίνωση των ε, ε, υδροφόρων οριζόντων και την, ε, των αρδεύσεων γύρω από το φυσικό δρυμό Δονιάνα. Αυτά θα κάνουμε. Θα στείλουμε και επιστολή και στον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ισπανικής Κυβερνήσεως και θα ζητήσουμε να εξετάσει και την αξιολόγηση των σεισμικών κινδύνων του έργου. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα και βεβαίως θα τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας καθώς και καλή επάνωδο στις αιστείες σας. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι στην χώρα σας. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή όρεξη και θα τα ξαναπούμε στις 2.30.